<coughs> Αρχίζουμε αγαπητοί συνάδελφοι. Good morning. Η πρόεδρος λέει καλημέρα. Αρχίζουμε. Καθίστε παρακαλώ. Comenzamos. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Ναι, μισό λεπτό. Ξεκινάμε. Ξεκινάμε. Σε όλους και όλες καλημέρα. Ξεκινάμε λοιπόν τη σημερινή συνάντησή μας. Έχουμε το πρώτο σημείο της ημερησίας διάταξης, η υιοθέτηση αυτής. Αν συμφωνείτε να σας πω ότι θα εντάξουμε στις ψηφοφορίες από τη στιγμή που έχουν συμφωνήσει όλες οι ομάδες το gender mainstreaming στην στρατηγική του 2020 έχουν συμφωνήσει όλες οι ομάδες, άρα λοιπόν θα μπορούσε να ενταχθεί και η ψηφοφορία αυτή στην ημερήσια μας διάταξη. Τι έχω να σας πω εγώ. Δύο πράγματα. Η Επιτροπή μας ε, που είχαμε τις 6 Οκτωβρίου ματαιώνεται γιατί θα έχουμε τις ακροάσεις των Επιτρόπων ε, και το καταλαβαίνουμε ότι αρκετοί από εμά και από εσά θα πρέπει να συμμετάσχουμε σε αυτές τις ακροάσεις. αλλά λοιπόν από τη στιγμή που δεν είχαμε κατεπήγοντα θέματα στη μέση μας διάταξη, τότε ε, ματαιώνεται η Επιτροπή μας. Να σας πω επίσης και κάτι άλλο. Θα θέλαμε να καλωσορίσουμε μία ομάδα επισκεπτών από το Μαρόκο. Δύο νεαρές ε, που σκηνοθετούν μία ταινία κινηματογραφική. Δεν ξέρω αν θα προφέρω καλά. Χάουνταλακουχάρ. Αν Μασάν Χατσάρι, δεν ξέρω αν πρόφερα καλά τα ονόματά τους, χαιρόμαστε που είναι εδώ μαζί μας. Δύο σκηνοθέτησες λοιπόν και από ό,τι είχαμε πει και μαζί τους ε, τους είχα πει ότι χαιρόμαστε που τις βλέπουμε εδώ από παντού από τον κόσμο και εκτός Ευρώπης να έχουμε γυναίκες που δίνουν τη μάχη τους για την ισότητα και σε τομείς, σε κλάδους που χρειάζεται κάτι παρόμοιο. Θα ήθελα να τις καλωσορίσω και να τις προσκαλέσω να ακούσουν τα σαν θα λεχθούν εδώ και θα προβληθεί στη μία το μεσημέρι η ταινία που έχουν γυρίσει και που έχουν σκηνοθετήσει και είστε όλοι καλεσμένοι για να την δείτε. Eh, λοιπόν, για τη συνάντηση τώρα των συντονιστών ε, που είχαμε να σας πω ότι καταφέραμε και τελειώσαμε το πρόγραμμα εργασίας για το 2015 με διάφορες ακροάσεις, χθες πρωτοβουλίες και αυτές οι συμφωνίες ε, τις οποίες κλείσαμε θα, θα ενημερωθείτε για αυτές και η Διεθνής Μέρα της Γυναίκας ε, για το 2015 το κύριο σημείο εργασίας εκεί και συζήτησης θα είναι το θέμα με το πώς θα ενισχυθούν οι γυναίκες και τα νερά κορίτσια μέσω της ε, μόρφωσης εκπαίδευσης. Αυτό λοιπόν για την Διεθνή ημέρα γυναίκας του 2015. Πάμε στο επόμενο σημείο. Η έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης μας συνάντησης ε, έλαβε χώρα στις 7 Ιουλίου. Και πριν να ψηφίσουμε, η κυρία Κορατσαβίντ επιθυμεί το λόγο. Ευχαριστώ. Σύντομα κύριε Πρόεδρε, ήθελα να σας πω ότι πολλές από εμάς Πάμε από τη μία επιτροπή στην άλλη. Και όταν υπάρχει ψηφοφορία, το να περιμένουμε 20 λεπτά, δείχνει έλλειψη σεβασμού. Οπότε παρακαλώ. Αφού έχουμε ψηφοφορία, όσα σημαντικά και να έχουν οι συντονιστέ, θα έπρεπε να μπορούμε να κάνουμε ψηφοφορία όταν προβλέπεται. Por supuesto, la próxima πρώτη, την φορά σίγουρα θα το προσπαθήσουμε αυτό, αλλά ζητάω την κατανόησή σας. Εδώ ξεκινάμε τη νέα θητεία. Έχουμε δουλειά και συντονιστές παντού και η πρόεδρός σας. Και ακριβώς θα πρέπει σιγά σιγά να προσαρμοστούμε και αυτό μας προκαλεί δυσκολίες πολλές φορές. Εντάξει, και θα σας ευχαριστώ πάντως για την υπομονή σας και για την ε, διάθεσή σας ε, συμμετείχατε και συντονίστριες και έτσι μπορέσαμε μέσα από ένα διάλογο και συμφωνίες να καταλήξουμε για, να ληφθούν κατά πλειοψηφία απόφαση. Πολλές φορές απαιτεί περισσότερο χρόνο. Πάντως θα το προσπαθήσουμε αυτό την επόμενη φορά να είμαστε ταχύτεροι και να σεβαστούμε την ώρα. Να ψηφίσουμε τώρα.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 abstenciones aprobado enmienda número 3 votos a favor votos en Τρία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Προχωράμε. Ψηφίζουμε τις τροπολογίες για τη στρατηγική του 2020. Οκτώ οι τροπολογίες. Όλες μαζί αν θέλετε. Εκτός αν κάποια ομάδα θα ήθελε να τις ψηφίσουμε ξεχωριστά. Όλες μαζί. Ναι. Ναι. Μία ως οκτώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. εγκρίνονται. Εγκρίνοντες. Ευχαριστώ. Εδώ σχετικά με τις ακροάσεις κάτι ενημερωτικά. Στην διάσκεψη των Προέδρων είχε αποφασιστεί ότι στην περίπτωση αυτή σχετικά με την εξέλιξη, τι θα γίνει με τις ακροάσεις. Εδώ αλλάζουν τα πράγματα σχέση με άλλες φορές ε, που κάθε φορά σε κάθε επιτροπή διαπραγματευόταν κανείς τι έγινε, τις ερωτήσεις κλπ. Αλλά ξε... αλλάζει τώρα η μέθοδος. Σε κάθε ακρόαση δίνουμε χρόνο για κάθε πολιτική ομάδα και σε κάθε πολιτική ομάδα εκεί θα πρέπει να ρυθμιστεί το τι ερωτήσεις, πόσο χρόνο θα διαρκέσουν κλπ. για τις επιτροπές ε, με τις ακροάσεις αυτές. Η βασική για μας ακρόαση είναι της κυρίας Γιουρόβα. Μαζί με την Ίνκο, τη Λίβε και την ε, νομικών υποθέσεων και καθένας από τους συντονιστές συντονίστριε, όποιου μπορούμε θα διαπραγματευτούμε ακριβώ πόσο χρόνο θα έχουμε στη διάθεσή μα για να υποβάλουμε ερωτήσει σχετικά με αυτά τα θέματα για την ισότητα στην κυρία Γιούροβα. Στη συνάντηση των συντονιστών τη συμφωνήσαμε για τα σημαντικότερα θέματα αυτά να τεθούν επιτάπητος και κάθε φορά που ο συντονίστης γνωρίζει πόσες θα είναι αυτές οι ερωτήσεις, πώς θα διαρκέσουν λοιπά για την ισότητα, τότε να τα έχουμε αυτά στα χέρια μας για να μην ε, ακουστούν πέντε ερωτήσεις ας πούμε για το ΠΕΓΑΠ και καμία άλλη για τη βία ανάμεσα στα φύλλα. Δηλαδή, να ξέρουμε τι θα ρωτήσουν και οι υπόλοιποι, ώστε να μην έχουμε επικάλυψη ερωτήσεων. Αυτό. Και επειδή συμμετέχουμε ε, και στην ακρόαση της κυρίας Τάισον σχετικά με την, ε, και με την Επιτροπή απασχόλησης κοινωνικών υποθέσεων και αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι να έχουμε την εγγύηση ότι λίγο πολύ όσος θα έχει την Προεδρία εκεί να μπορέσει να ε, υποβάλει ένα-δύο ερωτήσεις και αυτό είχαμε πει και από τις διάφορες ομάδες να μπορέσουμε να καλύψουμε το θέμα αυτό. Επειδή ρωτήθηκε, μέχρι τώρα δεν είχαμε σαφή απάντηση ποιες θα είναι οι αρμοδιότητες ε, ανάμεσα σε αυτές τις δύο επιτρόπους για την αναθεώρηση της οδηγίας, ας πούμε, για θέματα μητρότητας. Δεν ξέρουμε η κυρία Γιώροβα θα είναι ή η κυρία Τάισον η υπεύθυνη, η υπευθυνη αρμοδια Δεν το ξέρουμε αυτό μέχρι τώρα και ελπίζουμε μια κάποια στιγμή και μάλιστα σύντομα να το γνωρίζουμε ώστε να ξέρουμε ποιαν θα ρωτήσουμε τι. Ε, αυτά που θα ρωτήσουμε να αντιστοιχούν ε, σε αυτά που θα έχει σαν καθήκοντα. Αυτά ήθελα λοιπόν να σας πω ενημερωτικά. Δεν ξέρω τώρα μήπως... Ποιος άλλος, η κυρία Μορμπάη, έχει ζητήσει το λόγο. Yes, uh, thank you very much. Uh, as I understand... Uh, σας ευχαριστώ πολύ. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ε, αποφάσισε για τη συνάντηση των συντονιστών σε σχέση με την επισκόπηση που θα πρέπει να δίδεται εγγράφω σε όλα τα μέλη. Να αποτυπώνεται δηλαδή γραπτά το θέμα και η συζήτηση των συντονιστών. Ένας από τους λόγους είναι ότι εμείς είμαστε μη εγγεγραμμένοι Βουλευτέ, δεν ανήκουμε σε οποιαδήποτε ομάδα, αλλά έχουμε πλήρη δικαιώματα και εμεί θέλουμε λοιπόν να ενημερωνόμαστε. Και στο πνεύμα λοιπόν αυτό θα ήθελα να σα ερωτήσω κατά πόσον σύμφωνα με τις αρχές της δικαιοσύνης και της αναλογικότητας θα έχω την ευκαιρία να θέσω ερωτήσεις. Ελπίζω να θεωρείτε ότι έχω τα επαγγελματικά προσόντα. Ήμουν και μέλος επί τέσσερα χρόνια ε, της Επιτροπής ΣΥΤΟ στα Ηνωμένα Έθνη. Ελπίζω λοιπόν να έχω την ευκαιρία να θέσω και εγώ ερωτήσεις. Ναι, σχετικά με το πρώτο θέμα. Όταν αναγγείλαμε τα αποτελέσματα για την συνάντηση των συντονιστών, σας είχα πει ότι Για όλες αυτές τις υποθέσεις που ασχοληθήκαμε για τις συμφωνίες, οι σχετικές πληροφορίες θα δοθούν σε όλους τους συναδέλφους, όλους τις συναδέλφισες εδώ. λοιπόν, για να ενημερωθούμε για τις αποφάσεις. Σχετικά με τις ακροάσεις τώρα. Αυτό που μου λέει η γραμματεία είναι ότι υπήρξε μια συμφωνία σε κάθε μία από αυτές τις ακροάσεις οι μη εγγεγραμμένοι επίσης θα μπορέσουν να επιβάλλουν δύο ερωτήσεις ε, γι' αυτό. Μήπως ε, θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε με τις μη εγγεγραμμένους για να δούμε ποιες θα είναι αυτές οι ερωτήσεις τους και ποιος θα τις υποβάλει. Και οι υπόλοιποι θα διαπραγματευτούμε με τις ομάδες μας για τις ερωτήσεις ε, και το ίδιο και στις επιτροπές σα επαναλαμβάνω για να υπάρχει δυνατότητα, υπάρχει δυνατότητα αυτή για τις δύο ερωτήσει. Αυτά και πολύ καλά. Κανείς άλλος δεν θέλει να ρωτήσει κάτι. Το επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης έχει να κάνει με την έκθεση για την ισότητα ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες για την έκθεση αυτή του 2013. Ο κ. Ταραμπέλα, εισηγητής πρώτη ανταλλαγή απόψεων σήμερα χωρίς όμως κανένα έγγραφο για να ακούσουμε τις διάφορες απόψεις των συναδέλφων σχετικά και έτσι ο εισήγητης να μπορέσει να ξεκινήσει με ένα πρώτο προσχέδιο. Ξέρετε, έχει αιτήσιο χαρακτήρα αυτή η έκθεση και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να κάνει μια εκτίμηση τι γίνεται, πώς, προχωρούν, πώς προχωράει αυτή η πολιτική εξαφάνιση των ενισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών. Είναι σημαντική η έκθεση γιατί χρησιμεύει. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα έτοιμο πολιτικό προς ποια πολιτική θέλουμε να στραφούμε, να υπάρξουν βήματα, να κατευθυνθούν προσπάθειες, να ζητήσουμε από τα διάφορα θεσμικά όργανα, να προσέξουν ιδιαίτερα την ανάπτυξη αυτών των πολιτικών και θεωρώ ότι ελπίζω σε αυτήν την πρώτη συζήτησή μας να μπορέσει να ωφελήσει αυτή η συζήτηση ο Σταραμπέλα να βοηθεί ο ίδιος στην εργασία του και στην έκθεση αυτή να μπορέσουμε να λάβουμε, να λάβουμε μια θέση σε βασικές πολιτικές στην εργασία μας σαν κοινοβούλιο. Ο κύριος Ταραμπέλα έχει το λόγο λοιπόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι, χαίρομαι ιδιαίτερα. Με τιμάει το ότι ορίστηκα εισηγητής για την έκθεση αυτή. Εδώ στο ξεκίνημα της θητείας Είχα την ευκαιρία ήδη την ίδια εργασία να κάνω το 2009-2010 στο ξεκίνημα επίσης ε, της προηγούμενης θητείας και στο τέλος ε, απορρίφθηκε μια έκθεση. Αυτό έγινε δυστυχώς μόνο στο τέλος της θητείας μας. Αυτό θα πρέπει να το αποφύγουμε. Γι' αυτό τώρα ξεκινώντας, εντάξει όχι να χρησιμοποιήσω πάρα πολύ χρόνο, αλλά κάποιο χρόνο έχουμε πολλούς νέους συναδέλφους ε, και να συνεργαστούν με το σκιώδη συγητή και οι περισσότεροι συμμετέχουν ε, σε δύο, τρεις και τέσσερις ε, επιτροπές και χρειάζεται να δούμε πώς θα υπάρξει μια συνένεση και θα επανέλθω λοιπόν να ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος μας τα σημαντικά θέματα σχετικά με την εξέλιξη αυτή της ισότητας ή τη μείωση των ανισοτήτων, για να το πω καλύτερα. Έχουμε 7 θέματα που θα πρέπει να εξτάσουμε κάτι την απόψή μου. Το πρώτο σχετικά με την κρίση, αυτή συνεχίζεται λοιπά, Δεν έχουμε μια ανάκαμψη στην Ευρώπη και όλα αυτά επηρεάζουν ιδιαίτερα τη γυναίκα και τις συνθήκες εργασίας της και η μερική απασχόληση και αυτή επηρεάζει ιδιαίτερα εδώ τα πράγματα και οικονομικά και το να μπορέσει κανείς να απασχοληθεί πλήρω, αυτό είναι κάποιος δύσκολο και επίσης για τους στόχους της Βαρκελόνης το 2002 και για να το πετύχαμε θέλαμε το 2010 δεν τα καταφέραμε σχετικά με την ποιος φυλάει τα παιδιά, ποιος έχει τα παιδιά και βλέπουμε ότι επιβαρύνει τη γυναίκα και πώς θα μπορέσει να συνδυάσει, να συμφιλιώσει την επαγγελματική με την οικογενειακή της ζωή. Σημαντικό είναι αυτό. Θα πρέπει να δούμε επίσης για την ε, φορολογία. Δεν έχουμε και αρμοδιότητες, είναι των κρατών μελών, αλλά ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη σίγουρα θα πρέπει να προχωρήσουν σε μία ανάλυση αυτή σε αυτής της φόρων σε αυτόν τον κόσμο, γιατί σαν εργαλείο είναι εις βάρος των γυναικών που εργάζονται. Για να δούμε λοιπόν πώς τα πράγματα θα μπορούσαν εκεί να βελτιωθούν. Τέταρτο σημείο. Αυτά που είπε η Επιτροπή στο ξεκίνημα ήταν πολύ θετικά. Ίσως από εκεί θα πρέπει να ξεκινήσω. Τιμώντας τα και μια κάποια... κάνω κάποια παραπονό αυτή τη μητρική άδεια δεν την λεθεί ιδιαίτερα και είχε μείνει κάπως στο ψυγείο μέχρι να ληφθεί απόφαση από το Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο και ίσα ίσα που είχε περάσει θέση το Κοινοβουλίου με δύο αντίθετα στρατόπεδα κάπως η κυρία Μωρέτ ε, και με τον σκιώδη συγητή αλλά θα έπρεπε να το βγάλουμε από το ντουλάπι αυτό στην και αυτό το pay gap, αυτές τις διαφορές ε, μισθού αμοιβή ε, είναι 16 με 20% από ό,τι υπολογίζεται. Αλλά αν ακολουθήσουμε αυτό το ρυθμό, ε, τότε σε μερικές δεκάδες χρόνια τα ίδια θα λέμε πάλι. Εντάξει, μια κάποια πρόοδος επιτυχάνεται, αλλά παρατηρείται πάντα μια ανισότητα όσον αφορά τις αμοιβέ και είναι αδικία εις βάρος των γυναικών. Το επόμενο σημείο είναι η βία κατά των γυναικών και ζητάμε εδώ και αρκετά χρόνια πώς θα ε, θεσπιστεί μια χρονιά κατά της βίας ε, κατά των γυναικών. Δεν το είδαμε ακόμα να γίνεται και εδώ είχαμε τώρα μια δήλωση κάτι το συμβολικό. Δεν είχαμε καμία δυνατότητα θα χρειαζόταν κανονικά να είχαμε πολλές περισσότερες υπογραφές. Θα ήταν και κάτι το συμβολικό, αλλά κυρίως ε, μέσω του ίντερνετ ε, η βία. Δεν είναι μόνο φυσική, είναι ηθική, ψυχολογική και πολλές γυναίκες υποφέρουν ας πούμε. Μια κοπέλα 16, ένα κορίτσι 16 ετών ε, αυτοκτόνησε γιατί την παρενοχλούσαν μέσω του ίντερνετ. Έπαιρνε τόσα πολλά και άσχημα μηνύματα και καταλαβαίνετε. Άρα λοιπόν υπάρχει και αυτή η κυβερνοβία. Αυτό το επόμενο σημείο το έβδομο είναι το πώς ε, κάθε γυναίκα στην Ευρώπη θα μπορούσε ε, να διαθέσει το σώμα της όπως θέλει για την άβλωση, για την αντισύλληψη, το ίδιο υποστήριζω προς το 2009 και η παράγραφος αυτή είχε ψηφιστεί ε, με ιδιαίτερη πλειοψηφία. Ε, χρειαζόταν όμως να το πω ολοκλήρωσα. Ίσως επίσης να δούμε και το πρόβλημα, έχουμε κι άλλο, πως τη φτώχεια ας πούμε, τη φτώχεια σχετικά με τις μονογονικές οικογένειες, ε, που τις γυναίκες μόνες πολύ συχνά, να δούμε αυτό το Ταμείο Εγγύησης για την ε, ότι νεολαία που είναι σημαντικό εργαλείο ανάκαμψης, σημαντικό είναι επίσης τα νικητικά συμβούλια, οι ποσοστώσεις γυναικών, θα τα δούμε αυτά τα πράγματα, αλλά το είπα και στους συναδέλφους από την παλιά θητεία του Κοινοβουλίου και στους νέου, μερικές φορές επειδή βάζαν πάρα πολλές λεπτομέρειες στην ετολική σκέψη, σε πολλέ παραγράφους εδώ και εκεί, ε, σε παραγράφους που καμιά φορά και δεν χρειαζόταν συσσαγωγικά. Ε, σε αυτά που πρέπει όλοι μας να υπερασπιστούμε. Γι' αυτό κάπως ε, να απαλλαχτούμε από διάφορες σκέψεις που από ό,τι είδαμε αυτή η απόρριψη ήταν ιδιαίτερα νοτική ένδειξη και ε, ακριβώ το έριξαν στα σκουπίδια γιατί υπήρχαν πολλά και διάφορα εκεί που τα θίγαμε υπερβολικά, που υπήρχαν αντιφάσει των ατάλλων. Αυτά λοιπόν ένα βασικό θεμελιώδης κείμενο που να λέει ποια τα βασιλευτικά δικαιώματα και υπολογίζω στην βοήθειά σας κυρία Πρόεδρε και είμαι όλος αυτιά για να σας ακούσω, να ακούσω την άποψη του καθένα σας. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ κύριε Ταραμπέλα για την εισήγησή σας και τώρα ας αρχίσει ένας γύρος τραπέζι, μια συζήτηση και ξεκινά πρώτη η κυρία Νόελ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλή αυτή έκθεση. Νομίζω ότι η έκθεση περιλαμβάνει πάρα πολλούς ε, σημαντικούς τομείς. Θα ήθελα όμως να προσθέσω άλλο ένα πολύ σημαντικό θέμα σε ό,τι αφορά την κακή πολιτική, την υγειονομική πολιτική. Επανειλημμένα εμφανίζεται το πρόβλημα αυτό. Οι δοκιμές για τα φάρμακα και οι υποσολογίες και η χρήση των φαρμάκων βασίζονται πάρα πολύ και υπερβολικά μη αναλογικά, δυσανάλογα στο σώμα των ανδρών. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό και αφορά και την ιατρική ευθύνη που υπάρχει τα θέματα αυτά, γιατί φυσικά είναι επιζήμιο για τι γυναίκε. Τονίζω λοιπόν και το τομέα αυτόν. Ε, ε, Ευχαριστώ. Επόμενη, η κυρία Μορβάη. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με προσοχή άκουσα τον κύριο Τραμπέλα, πάντα μεγάλα μου χαρά είναι αυτή. Όταν ένας άντρας ε, μιλάει για θέματα ισότητας γυναικών και ανδρών και τάσεται υπέρ αυτών. Αλλά είναι σημαντικό λοιπόν το γεγονός ότι οι, γυναί... Ε, οι άντρες τάσσονται υπέρ του δικαιώματος στην άμβλωση. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στους άντρες συναδέλφους ότι δεν τίθεται θέμα πραγματικής ε, ελεύθερης επιλογής στην πραγματικότητα. Καμία γυναίκα δεν αποδέχεται ευχαρίστως την άμβλωση. Στις περισσότερες περιπτώσεις εξαναγκάζεται. Και αυτός ο εξαναγκασμός προέρχεται ε, συχνά από τους άντρες, από τον ίδιο τον άντρα συχνά της κάθε γυναίκας. Αλλά και σε πολλές περιπτώσεις η γυναίκα έχει άλλη άποψη για το μαρτύριο της ε, άμβλωσης. Και αυτό γιατί ο σύντροφός της ενδεχομένως να μην έχει τη διάθεση να αναλάβει το, την ευθύνη του. Και αυτό λοιπόν ε, συνδέεται με την ε, ψυχική βία, με τον πόνο της αφαίρεσης του παιδιού της. Θα πρέπει να φροντίσουμε λοιπόν οι άντρες πιο ενεργά να υποστηρίζουν τις γυναίκες, προκειμένου να μπορούν συνήθως, γιατί όταν μιλάμε για αναπαραγωγικά δικαιώματα, αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο εφόσον οι άντρες ε, εκπληρούν τα καθήκοντά τους. και όχι απλά να περιορίζονται στη γονιμοποίηση. Να παρακαλέσω λοιπόν τον κύριο Ταραμπέλα και τους ε, άνδρες συναδέλφους του να φροντίσουν προκειμένου να πιστούν οι άνδρες ότι υπάρχει ευθύνη και από πλευρά του άνδρα. Και όταν έχει συμβεί η εγκυμοσύνη να αναλαμβάνουν τις, τα καθήκοντά τους, τις υποχρεώσεις τους και όχι μόνο να τα κοιτάνε αυτά ως ε, υποχρέωση των ανδρών. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα έχει το λόγο ο κύριος Ουκάτσον. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Ταραμπέλα για την παρουσίασή του. Μου άρεσε πώς τα παρουσιάσατε, ποια θίξατε σαν σημεία. Να επιμείνω σε ορισμένα σημεία που θεωρώ σημαντικά να προσπαθήσουμε να επιμείνουμε στην φετινή έκθεση στο πώς ε, οι διδακτικές μεταρρυθμίσεις επηρεάζουν την κατάσταση στο θέμα αυτό. Νομίζω ότι επηρεάζουν πολλά και ιδιαίτερα μάλιστα τα εργασία της ε, συντάξει, τα ηλικιωμένα άτομα στη φάση αυτή. Σημαντικό λοιπόν θα είναι στην έκθεση να μπορέσουμε να εστιάσουμε ιδιαίτερα πάνω στα σημεία αυτά και το είπατε επίσης ε, σαφώς το θέμα της βίας όλους μας αφορά και θα πρέπει να κάνουμε μια σύντομη ανάλυση πώς οι περικοπές στον προπολογισμό για το θέμα επηρεάζουν την κατάσταση γιατί υπάρχει μια αύξηση της βίας ε, σε διάφορες χώρες. Εντάξει, ίσχυε αυτό αλλά πάμε από το κακό στο χειρότερο στις χώρες αυτές. Ενισχύεται το φαινόμενο και στην έκθεση θα πρέπει να επιμείνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Επιτροπή χρειάζεται να υποβάλει πρόταση για οδηγία, δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Να επιμείνω λοιπόν και σε αυτό. Σύντομα τρία σημεία ακόμα. Για τη φτώχεια, το είπατε. Έχει να κάνει με τα ηλικιωμένα άτομα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό και επίσης παρουσία γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Σημαντικό και αυτό πρέπει να το εξετάσουμε και κάτι ακόμα. Ήταν το έβδομο σημείο σας. Χρειάζεται στην έκθεση να μιλούμε για το πώς η γυναίκα θα πρέπει να διαθέτει όπως θέλει το σώμα της. Εντάξει, ε, δεν γίνεται να μην επιμείνουμε στο σημείο αυτό από τη στιγμή που λαμβάνουμε απόψη μας τι γίνεται σε διάφορες χώρες. Η Ισπανική κυβέρνηση επιτέλους απέσυρε το νέο νόμο για τις αμβλώσεις χθε, αλλά έχουμε παντού διαρκείς επιθέσεις και κινδύνους. Θα πρέπει να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα πάνω στο θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Sí, muchas, muchas. Σας ευχαριστώ πολύ. Υποστηρίζω καταρχήν και καταρχάς ε, κάτι που θα μπορούσε να είναι θετικό και να μην καταλήξει όπως πέρυσι που την τελευταία στιγμή απορρίφθηκε από το Κοινοβούλιο η έκθεση και δώσαμε μια εικόνα ιδιαίτερα αρνητική στους Ευρωπαίους πολίτες αλλά και στις Ευρωπαίες γυναίκες που άλλα έλπιζαν. Ελπίζομαι να σταθούμε στο ύψος των απαιτήσεων φέτος και να δείξουμε ότι είμαστε υπεύθυνοι πολιτικοί. Συμφωνώ με τα σημεία που πρόβαλε ο εισηγητής Ρίχνοντας μια ματιά στην έκθεση της Επιτροπής, ε, ακόμα μια χρονιά βλέπω, διαπιστώνω ότι θριαμβεύει η ανισότητα παντού και στην εργασία και εντάξει κρίση, βία, στα διοικητικά συμβούλια. Με την έκθεση αυτή που θα επεξεργαστούμε όμως θα πρέπει να προχωρήσουμε ένα βήμα ακόμα. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να προωθήσουμε μια ακόμα οδηγία σχετικά με τις εκθέσεις, με, τις, ε, με τη μετρική, με τη γονική άδεια, μητρική, υπατρική, με την παρουσία και λοιπά στα διοικητικά συμβούλια και εδώ για τη βία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να λάβουμε υπόψη μας ε, την πρώτη έκθεση που είχε συνταχθεί σχετικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει όπως σας είπα να προσφέρουμε το κάτι παραπάνω Εκτός από την άλλη διάγνωση αυτής της δύσκολης περίπτωσης, ε, να υποβάλω μια πρόταση. Τι θέλουμε να κάνουμε με την έκθεση αυτή. Τουλάχιστον να δούμε ποιες είναι αρμοδιότητές μας σαν κοινοβούλιο και να επιμείνουμε να επηρεάσουμε τις προτεραιότητες. Αυτό θα πρέπει να κάνουμε σε αυτή τη θητεία του Κοινοβουλίου. Μια οδηγία για τη βία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ναι, Έχουμε ευρωπαϊκά κράτη που θεωρούν ότι είναι ιδιωτικής φύσεως θέμα η βία. Απαράδεκτο. Δεν έχουμε αριθμούς και στατιστικές, μόνο μια έρευνα που έδειξε όμως και καθαρά τις επιπτώσεις της βίας στην Ευρώπη κατά των γυναικών. Θα πρέπει να δούμε επίσης βέβαια και τη φτώχεια πώς επηρεάζει. Αυτές τις διαγνώσεις όμως τις βλέπουμε κάθε χρόνο. Θα πρέπει να δούμε τις προτεραιότητες εδώ μέχρι το τέλος να δούμε τις οδηγίες για τα διοικητικά συμβούλια, μια συνοχή, εργαλεία εναρμονισμένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο με συστήματα κατάλληλα για να μπορέσουμε έτσι να κάνουμε μία σύγκριση στοιχείων επίσης σε κάθε ε, τομέα, σε, όλα τα κράτη, να δούμε τις βέλτιστες πρακτικές, ε, να δούμε γιατί σε μερικά κράτη έχουμε θετικά αποτελέσματα και άλλοι όχι και να προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε. Εφορετικά το να κάνουμε διαγνώσεις, να βλέπουμε αριθμούς, όλα αυτά επαναλαμβάνονται συνεχώς. Δεν πρόκειται για ένα βήμα προς τα εμπρός, αλλά θα πρέπει να το κάνουμε αυτό το βήμα για το μέλλον. Θα ήθελα λοιπόν στην εργασία αυτή, για την έκθεση αυτή, να ε, επικεντρώσουμε την προσοχή μας στα θέματα που είπα. Ευχαριστώ. Och Σας ευχαριστώ. Και έχω ασχοληθεί όπως ο κ. Ταραμπέλα έχω ασχοληθεί αρκετό καιρό και θέλω να δω τι θα γίνει όσον αφορά τελικά την υπόθεση αυτή και γιατί πέρσι δεν τα πήγαμε καλά όταν ήρθε η ώρα του να ολοκληρώσουμε το έργο μας γιατί σε αυτά τα ζητήματα έχουμε κάποιο πίσω γύρισμα και βέβαια πολλές είναι γυναίκες που έχουν πληγεί από αυτή την ε, οπισθοδρόμηση με ναι. ταράζει πάρα πολύ όταν βλέπω ε, τι γίνεται τη μία χρονιά μετά την άλλη. Είναι πολύ σημαντικά τα θέματα αυτά. Θα πρέπει σε κάθε κράτος μέλος, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση να τα αντιμετωπίσουμε. Θα πρέπει να προχωρήσουμε θαραλέα. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση και όσον αφορά την ίσια αμοιβή για δουλειά και το θέμα της γονικής άδεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορεί κανείς να έχει το δικαίωμα κανείς να κάτσει σπίτι με τα παιδιά του και οι άντρε και οι γυναίκες. Μέχρι ότου το καταφέρουμε αυτό, τότε οι, μέχρι τότε οι άντρε θα μα καπελώνουν. Ο Μαρκίρ είπε για του ε, στόχου τη στόχους της ε, τι γίνεται για στην προσχολική περίοδο, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τους ε, ηλικιωμένους. Ε, και στη χώρα μου έχουν γίνει κάποια τέτοια βήματα λοιπόν ε, για να καλύψουν τους ηλικιωμένου και πάρα πολλές γυναίκες δουλεύουν part-time, μερική απασχόληση, για να κάτσουν σπίτι να φροντίσουν τους ηλικιωμένους. και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είτε πρόκειται για πεθερικά, είτε πρόκειται για αγωνίες, να μπορεί κανείς να τους φροντίσει. Ε, άλλωστε τώρα ο κόσμος ζει ε, περισσότερο χρόνο και βέβαια υπάρχει πρόβλημα και με τις συντάξεις. Τέλος, ε, όσον αφορά το εμπόριο ανθρώπων, το δουλεμπόριο, το 2011 θυμάμαι το συζητήσαμε. Διαπιστώσαμε τότε ότι υπάρχει αύξηση αυτού του δουλεμπόριου. Παρακαλώ και αυτό να το καλύψουμε και του χρόνου τα, τα πρόκειται να υποβάλουν εκθέσεις σε σχέση με το τι έχουν κάνει ε, για το πρόβλημα. Βεβαίω και συμφωνώ με τους συναδέλφους για όσα είπαν για τα προβλήματα τα σχετικά με την υγεία. Θυμάμαι από την ΚΟΕ ε, ε, η κυρία Σβέντσον έγραψε μια πάρα πολύ καλή έκθεση για το πώς έχουμε δεσμευτεί διακρίσεις και στον τομέα της υγείας. Πολύ σημαντικό και αυτό. Ευχαριστώ. η κυρία Μπερντερ. Κινδυνεύοντας να φορτώσω και άλλο τον κύριο Τραμπέλα θα καταντήσει να γράφει διδακτορικό στο τέλος. Αλλά όντως έχει πάρα πολλά θέματα που καλύπτει εδώ και συμφωνώ με τους περισσότερους που τοποθετήθηκαν πάντως. Το θέμα που εγώ θα ήθελα επίσης να καλύψουμε την έκθεση είναι η πρόσβαση στην δικαιοσύνη. Θεωρούμε ότι έχουμε ένα σύστημα δικαιοσύνη, αλλά πολλές φορές οι γυναίκες δεν μπορούν να προσφύγουν στην δικαιοσύνη. Για πολλούς λόγους. Δεν έχουν χρήματα. Ή κάποια πράγματα δικαιώματα δεν είναι τα ίδια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για άντρε και γυναίκε. Το ίδιο ισχύει για το δίκαιο διαζυγίου. Ε, Πολλέ φορέ ε, για κάποια μικροεγκλήματα οι γυναίκε φυλακίζονται ευκολότερα από τους άντρες. Ε, σε πολλές περιπτώσεις επομένως υπάρχει ανισότητα και το όλο ζήτημα της προσβασιμότητας στη δικαιοσύνη είναι ακριβώς μία από τις κεκριμένες ανισότητες που θα πρέπει να τις εξετάσουμε. Πάντως, επισημένω ιδίω τους ε, καινούριου συναδέλφους, γιατί για μένα είναι αυτή η δεύτερη θητεία, είπαμε ότι είπαμε ότι σε κάθε επιτροπή ένας αντιπρόεδρος θα είναι αρμόδιος να εξετάζει τις ε, ανισότητες που υπάρχουν στην ε, αρμοδιότητά του. Στην αρμοδιότητα της επιτροπής δηλαδή. Πολύ χρήσιμο αυτό νομίζω και έτσι να δούμε ποιοι στις ε, διάφορες επιτροπές είναι οι αρμόδιοι για αυτή την ανισότητα των φύλων. Να έρθουμε σε επαφή μαζί τους και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σωστό τρόπο να δούμε τι μπορεί να κάνει το Κοινοβούλιο, τι μπορεί να καταφέρει για να αποδοθεί δικαιοσύνη στι γυναίκε. Αν γι' αυτό λοιπόν καλυφθεί την έκθεση θα είναι χρήσιμο. Πρόεδρος. Κυρία Αλεγκρίπ. σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. η κυρία Μαρία Γκαμπριέλ που είναι ισχυώδη συγγήτρια, είναι απούσα και μιλώ εκ μέρους της. Ε, και κανονικά εκείνη η συνομιλήτρια του κύριου Ταραμπέλα, τον οποίο θα ευχαριστήσω για την παρουσίασή του. Ήταν ιδιαίτερα σημαντική η παρουσίαση, την άκουσα πολύ προσεκτικά τα κύρια θέματα, τους τίτλους των κεφαλαίων, τους 7 πυλώνες σχετικά με την εκθεσή του. Θα τον ευχαριστήσω επίσης γιατί σίγουρα ε, διδάχτηκε από την αποτυχία της τελευταίας έκθεσης για τις ευκαιρίες ανάμεσα σε γυναίκες και άνδρες ε, της προηγούμενη θητεία και κατά την απόψή μου τα λόγια του ήταν ιδιαίτερα σοφά ε, για το για ποιους λόγους καταλήξαμε σε αυτή την αποτυχία. Υπήρχαν ορισμένε υπερβολικά προχωρημένες θέσεις και λοιπά και αυτά θα πρέπει λοιπόν να ενθαρρύνουμε για επόμενο χρονικό διάστημα να είμαστε λογικοί και με τον εαυτό μας και να μπορέσουμε να ενεργήσουμε όλοι μαζί επικοδοματικά από κοινού και είπε ο κύριος Τραμπέλα ότι θα συνεργαστεί με όλους, έστω και αν απαιτήσει χρόνο αυτό, να πετύχει μια συνένεση. Αυτό και απόψή μου είναι θετικό για να μπορέσει να ξεπεράσει τα εμπόδια και έτσι να μην πέσει σε αυτές τις παγίδες, ε, πάνω σε αυτές τις δυσκολίες, τις στήρες. Ε, δεν θα προχωρήσω σε λεπτομέρειες κάθε θέματος ε, από την πλευρά του ΕΛΚ. Η Μαρία Γκαμπριέλ θα εργαστεί σχετικά με τις προτάσεις των γυναικών και υπάρχουν αρκετές προτεραιότητες από την ομάδα μας. Σίγουρα αυτά θα εμφανιστούν προπαρασκευαστικά αλλά θα ήθελα να θίξω ένα θέμα που μας απασχολούν και όλες ε, και στο ΕΛΚ σίγουρα αυτό μας έχει ιδιαίτερα ευαισθητοποιήσει και ανησυχήσει και κινητοποιήσει για την ε, βία κατά των γυναικών, ε, κατά οποιασδήποτε εκμετάλλευσης, κατά αυτού του σκλαβοπάζαρου ε, ξέρετε ότι υποφέρουν ιδιαίτερα οι γυναίκες, τα νέα κορίτσια και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω που το έθιξε καθαρά το θέμα αυτό. Ε, σίγουρα το προσέχουμε, προσέχουμε αυτό το θέμα, αυτή την παράγραφο, αυτό τον πυλώνα, θα τα προσέξουμε, θα υποβάλουμε προτάσεις και για την βία στην ε, κατοίκον αλλά και για, στον κυβερνοχώρο και στο ε, νήσι αμοιβή, επίσης διάφορες ανισότητες σχετικά με τις συντάξεις ε, και τα θέματα αυτά θα πρέπει να τα προσέξουμε σε αυτή την έκθεση ιδιαίτερα και σίγουρα είναι από τα σημεία που ιδιαίτερα μας απασχολούν στο ΕΛΚΑ. Ας μην μακρηγορήσω θα εργαστούμε να πετύχουμε συμφωνίες ε, για τα περισσότερα τουλάχιστον από τα θέματα αυτά που αναφέρθηκαν, τα περισσότερα επαναλαμβάνω και για μία πρόσβαση επίσης σε δυνατότητες ε, μόρφωσης, κατάρτισης, εκπαίδευσης, ε, οπουδήποτε σε κλάδους σε επαγγελματικούς παντού και ακαδημαϊκά και αυτά θα μπορούσαν να αναφερθούν καθαρά επίσης με στην έκθεση που είναι τα όρια και πώς αποκλείονται από διάφορες δραστηριότητες στα νέα κορίτσια θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ίσης πρόσβασης παντού σε όλους τους κλάδους από όλους άνδρες και γυναίκες. Αυτά θα πρέπει να φερθούν σε αυτήν την έκθεση. Αυτό λοιπόν και ολοκλήρωσα. Είναι νομίζω ιδιαίτερα επικοδομητικό το κλίμα και όλα αυτά είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Θα θέλαμε να ενθαρρύνουμε και εμείς τον εισηγητή μας. Ξέρουμε ότι σε αυτό το θέμα όπως και σε άλλα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην αρχή της επικουρικότητας η ομάδα μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Μαρκ Τραντέλα για την παρουσίασή του και το πόσο έχει στρατευμένος είναι για τα θέματα των γυναικών. Θα πρέπει να το πούμε. Είμαστε σε μια έκθεση, που ε, σε μια επιτροπή, περισσότεροι, τα περισσότερα μέλη είναι γυναίκες Λοιπόν, ε, πρόκειται για προστιθέμενη αξία και όχι σκέτη χαρά που βλέπουμε αυτή την προσπαθιά του για τις γυναίκες. Τον ευχαριστούμε για όσα μας είπε. Τον ευχαριστούμε επίσης για τους 7 πυλώνες θέματα που αναφέρθηκαν στα πλαίσια αυτής της έκθεσης. Σίγουρα θα μπορούσαν να συμπληρωθούν και με διάφορες άλλες ειδικότερε ανησυχίες αλλά θα πρέπει έτσι να λάβουμε υπόψη μας το σύνολο αυτών των 7 θεμάτων με τον ειδικό χαρακτήρα στον καθένα του και να καλύψουμε έτσι νομίζω αρκετά πλήρως το θέμα των ίσων δικαιωμάτων των γυναικών στις γυναίκες. Ανάγνωση ιδιαίτερα σημαντική επίσης για την έκθεση αυτή είναι ότι η ανάγνωση αυτή γίνεται στα πλαίσια μιας κρίσης από το 2008, αυτή η οικονομική κρίση η οποία οδήγησε σε μια διαχείριση από ευρωπαϊκής πλευράς ε, για να μπορέσουμε να ελέγξουμε, να περιορίσουμε το δημοσιοέλλημα και σε κάθε κράτος έχουμε και σκληρότερες θέσεις, εντάξει και φορές όχι, και λιγότερο σχετικά με τη μείωση των δημοσίων δαπανών. Αυτές οι μείωσες δαπάνες ε, Υπάρχουν υπηρεσίες κανονικά που θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση γυναίκες για να βοηθηθούν. Είχαμε μιλήσει για την υγεία. Έχουν μια έκθεση τώρα που μας δείχνει ότι πάνω από 30% των γυναικών δεν έχει πρόσβαση ακριβώς αμέσως μετά τη γέννηση ενός παιδιού ή πριν από τη γέννηση. Δεν μπορούν να επισκεφθούν το γιατρό τους και να πάρουν τις σχετικές πληροφορίες όπως πρέπει. Είναι ευάλωτες λοιπόν αυτές οι γυναίκες επειδή δεν μπορούν να δοθούν οι απαραίτητες πρώτες πληροφορίες όπως πρέπει πριν και μετά τη γέννηση ενός παιδιού. Επειδή υπάρχει κρίση, ανέφερα το παράδειγμα αυτό, αλλά κάποιος είπε προηγουμένως και για τη μείωση των δαπανών όσον αφορά τα ηλικιωμένα άτομα. Όταν ε, το δημόσιο δεν οργανώνει όπως πρέπει την υποδοχή αυτών ηλικιωμένων ατόμων, το βάρος αυτό, μιλάω για βάρος, ε, μια γυναίκα θα πρέπει πέρα από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις να μπορέσει να βοηθήσει αυτό το άτομο το ηλικιωμένο. Ε, αυτό λοιπόν και στο μια ζωή στον ηλικιωμένο και θα έχει μια ζωή στον παιδιών ε, παντού είτε πρόκειται για παιδικούς σταθμούς, ε, ε για νηπιαγωγία κλπ. εδώ θα πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό για την ε, γυναίκα εδώ. Έχουμε την κρίση εδώ και πέντε χρόνια ασκούνται πολιτική ε, λιτότητας προϋπολογισμού, και θα πρέπει μια κάποια στιγμή να δούμε τα πράγματα και με το μάτι των γυναικών το τι όλα αυτά προκάλεσαν στο θέμα της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, τα αρνητικές επιπτώσεις. Σας ευχαριστώ. Κύριε Ζητνάσκα, εγώ θα ήθελα να σας επισύρω την προσοχή όσον αφορά το σημείο υπεριθμών 6 από όσα μας είπε η κυρία Ταραμπέλα. Εκεί δηλαδή που αναφερθήκατε στην βία και συγκεκριμένα γιατί ασχολούν πάρα πολύ με τους ε, αναπήρους και με τις μειονότητες των Ρωμά. Ε, έχω ασχοληθεί με το θέμα αυτό όσον αφορά τις κοινωνικές ομάδες που είναι οι πιο ευάλωτες στην βία. Και έχουμε δυστυχώς πολλές περιπτώσεις, ειδήσεις σε πολλές χώρες, όπου έχουμε κάποιες ανάπηρες γυναίκες, οι οποίες θα πρέπει να ε, αντιμετωπίσουν τη βία την οποία υφίστανται, πολλές φορές εξαρτώνται από αυτόν που τους επιτίθεται και στις κοινότητες των Ρωμά γίνεται το ίδιο και εκεί υπάρχει μεγάλη κακομεταχείριση συχνά, οπότε εάν έχουμε ως σκοπό να λύσουμε το πρόβλημα δεν αρκεί μόνο να γράφουμε τέτοιου είδους ε, ε, διατυπώσεις. Χρειάζεται κάτι να κάνουμε στην δε Σλοβακία η κατάσταση είναι μάλλον θλιβερή γιατί δεν έχουμε αρκετό χώρο για να καλύψουμε αυτές που υφίστανται την κακοποίηση. Δεν υπάρχει προσωπικό, αστυνομική, ε, για τις γυναίκες που βιάζονται ή τέλος που κακομεταχειρίζονται, οπότε θα πρέπει και στην ε, έκθεση να δούμε πώς έχει πραγματικότητα στις διάφορες χώρες. Θα πρέπει επομένω αυτό το οποίο θέλουμε να γίνει πραγματικότητα. Δηλαδή να βρεθεί κάποιο και να βοηθά τι γυναίκε που έχουν ανάγκη. Ευχαριστώ. Κύριε Μπιόρκ. Θα σα μιλήσω στα αγγλικά, λέει κυρία Μπιόρκ, γιατί έχω εδώ μια, ένα σημείο από την Βαλίνα, την Σκιώδη Συγήτρια, και θέλω να πει η κυρία Βαλίνα, ε, συμφωνεί με το περισσότερο που ήδη έχουν ακουστεί. Θα ήθελε η κυρία Βαλίνα να πει ότι αυτή η έκθεση ε, θα πρέπει να καλύψει και το ότι και η κρίση έχει το ρόλο της όσον αφορά τις ε, ηλικιωμένες γυναίκες, τις γυναίκες και την ε, φτώχεια κλπ. Αυτό να το λάβουμε υπόψη, οπότε ασχολούμεθα με το θέμα της ισότητας και τονίζει επίση και η Δεβαλίνα το τι γίνεται με την απασχόληση των γυναικών, γιατί έχουμε εδώ πέρα στοιχεία ποιοτικά και ποσοτικά στην αγορά εργασία. Έχουμε λένε και περισσότερου φραγμού για τι γυναίκε. Επίση και όσον αφορά τι συντάξει είναι 39% λιγότερο από όσο ε, οι άντρε. Ε, να δούμε τι θα γίνει με τις πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν όσον αφορά επομένως την είσοδο αλλά και η παραμονή των γυναικών στην νέα αγορά απασχόλησης. Θα πρέπει όλα αυτά να το προσέχουμε, τα είπαν οι προηγούμενοι, για να δούμε τι μπορεί να κάνει το κράτος ε, όσον αφορά τη λειτουργία του κράτους για να βοηθήσει στην ανεξαρτησία και την ισότητα. Επίσης, ε, λέμε εδώ ότι θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τη βία μεταξύ των φίλων σε όλε τι μορφέ και επίσης κύριε Βαλίνα συμφωνία όσον αφορά την πρόσβαση στην δικαιοσύνη. Είναι πάρα πολύ σημαντική υπόθεση. Επίσης προβληματίζεται όσον αφορά την επιρροή ε, κάποιων θεσμικών οργάνων από την Εκκλησία συνδεόμενους φορείς, όπου γίνεται στην Ισπανία και κάποια αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών. Πολύ σημαντική αυτή η εκθέση. Θα είναι ίσως η πρώτη έκθεση αυτής της ε, θητείας που θα πρέπει να έχουμε τέτοια ευρεία προσέγγιση. Mm, Καλημέρα σας. Να ευχαριστήσω και εγώ τον Μαρκ Ταραμπέλα για αυτή την έκθεση με τόσα συγκεκριμένα σημεία και για την προσέγγιση του μεθόδου την εργασία αυτή. Η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει διάφορα σημεία και νομίζω ότι είναι ανοιχτό απέναντι σε όλους μας. Να λάβουμε υπόψη μας ότι εδώ στις αίθουσες αυτές του Κοινοβουλίου και μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχουμε συνειδητοποιήσει ότι παίζουμε και ένα πολιτιστικό ρόλο. Αυτή η πολιτιστική διάσταση είναι και των ανδρών και των γυναικών. Διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και όλοι μας και όλες μας γνωρίζουμε, επειδή την πολιτική αυτή την έχουμε και σαν αποστολή και σαν εργασία, ότι τις μάχες για τις γυναίκες τις κερδίζουμε εάν μαζί μας έχουμε και γυναίκες αλλά και άνδρες. Και πάνω απ' όλα αν έχουμε κοντά μας την κοινωνία των πολιτών, χωρίς την οποία καμία πρόοδος. Και θα ήθελα να παρακαλέσω όλους να μην ε, περιορίζουν την πολιτική της γυναίκες μέσα σε κλειστούς ε, ιδεολογικούς χώρους. Αν λέμε ότι θα πρέπει να τα λύσουν τα γυναικεία προβλήματα γυναίκες, εγώ δεν είμαι μαζί σας, γιατί κοντά μου, δίπλα μου θέλω και γυναίκες και άνδρες ε, που να έχουν όραμα, που να καταλαβαίνουν, που να είναι ικανοί. Και δεν θα συμμετάσχω ακόμα και αν δω ότι για γυναικεία θέματα ε, ασχολούνται αποκλειστικά, επαναλαμβάνω, γυναίκες. Γι' αυτό ακριβώς επειδή κατανοήσαμε ότι η δική μας η αποστολή είναι πολιτιστική επίσης και θα ήθελα να εκφράσω την ανησυχία μου για το θέμα το μόρφωσης, κατάρτισης, εκπαίδευσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα η Επιτροπή αυτή θα πρέπει ξεκινώντας από αυτό το σημείο να τονίσει ότι χρειάζεται να ενισχυθεί το θέμα σχολείο. Οι δυνατότητες εκπαίδευσης οι ίδιες ίσες δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε εάν δεν έχουμε να ρίξουμε μια ματιά, ένα βλέμμα στο μέλλον, στις επόμενες γενιές και όχι να περιοριστούμε μόνο στα σημερινά προβλήματα, υπάρχουν τα προβλήματα, έχουμε το πολιτικό χρέος να τα επιλύσουμε τα προβλήματα αυτά, αλλά χρειάζεται να οικοδομήσουμε μια πολιτική ένωση αξιών, προθέσεων, ξεκινώντας από το σχολείο λοιπόν, θα πρέπει στην έκθεση αυτή και στην εργασία που θα επιτελέσουμε όλοι μας να υπάρξει και η διάσταση σχολείο εκπαίδευση. Και επίσης για την κυβερνοβία. Εδώ και με τις κοιόδες με είμαι έτοιμη να συνεργαστώ και να βοηθήσω και μέσω της εργασίας μας στην Ιταλία που υπάρχουν πολλές γυναίκες, κυρίως γυναίκες ε, τις οποίες βασανίζουν εισαγωγικά στο ίντερνετ και κάτω από αυτό το βάρος και την πίεση έχουμε και άσχημη κατάληξη πολλές φορές. Σχετικά με τη φτώχεια έχουμε το θέμα των συντάξεων που αφορά κυρίως τις γυναίκες. Είναι βαριά, είναι επιβαρυντική, είναι άσχημη, αρνητική ακριβώς επειδή σε πολλές περιπτώσεις εκείνες ε, αναγκάζονται να έχουν και άλλα βάρη, να μεγαλώσουν τα παιδιά και να βοηθήσουν και τα ηλικιωμένα άτομα, τους γονείς τους, πολλές φορές που χρειάζονται αυτή τη βοήθεια. Δεν θα ήθελα επιμείνω στη δική μου σαν εισηγήτρια προσπάθεια που καταβάλω, αλλά και αφορά όλους μας ε, το θέμα της ε, μητρότητας ε, χρειάζεται να υπάρξει μια κατάλληλη θέση γιατί αν κρατήσουμε μια άκαμπτη ιδεολογική στάση τότε το θέμα επίσης της άδειας μητρότητας δεν θα το πετύχουμε να το λύσουμε. Γι' αυτό μη γυρίζουμε γύρω γύρω. Θα πρέπει να δούμε τον στόχο μας, να δούμε πώς θα πετύχουμε αυτό που προσπαθούμε εδώ και χρόνια είτε θα το κάνουμε ιδεολογική σημαία, θα πετύχουμε τίποτα και δεν θα έχουν καμία αναγνώριση οι γυναίκες της Ευρώπης απέναντι σε εμάς. Εγώ θέλω αποτελέσματα. Αυτά θέλω να πετύχω εδώ. Είμαι και ασκοπολιτική για να πετύχω για κόσμο θετικά πράγματα και όχι προσωπική ικανοποίηση σε μένα. Αυτό λοιπόν και για την άδεια μητρότητας σε θέματα με επίσης πολιτιστικά, μια διαφορετική προσέγγιση, κατάλληλη να καταβάλουμε προσπάθεια ώστε από εδώ να ξεκινήσει το μήνυμα για τους γονείς, για μια συμφιλίωση το πώς θα συμμεριστούν το ρόλο τους οι δύο γονείς. Και εδώ είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε τη βοήθειά μας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, ε, Πετήρ. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να αναφέρω κάποια θέματα τα οποία έχουν ήδη αναφερθεί και θα ήθελα όμως παρόλα αυτά να τα εξετάσουμε. Μας απασχολεί το θέμα των ανθρώπινων ωραρίων στα άτομα που ασχολούνται στην παροχή υπηρεσιών. Ναι, ναι ιδιαίτερα των γυναικών, που εργάζονται τόσο πολύ χρόνο που δεν έχουν τελικά χρόνο για τις οικογένειές τους, για προσωπικό χρόνο και πολύ συχνά δεν πληρώνονται και επαρκώς. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται επηρεάζουν και την δημιουργία οικογενειών και τελικά αποτελούν κάτι το επιζήμιο για τις γυναίκες γιατί σήμερα η μητρότητα είναι ουσιαστικά ένα προϊόν πολυτέλειας. Δεν είναι δυνατόν να ισχύει αυτό λοιπόν. Θα πρέπει να εκτιμάται η συνεισφορά της γυναίκας στο σπίτι γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική η συνεισφορά της γυναίκας η οποία φροντίζει την οικογένεια με την ανατροφή των παιδιών και γι' αυτό λοιπόν Πιστεύω ότι και οι γυναίκες αλλά και οι άνδρες και οι μητέρες και οι πατέρες θα πρέπει να υποστηρίζονται και να μην γίνεται περικοπή στα μέσα αυτά. Το δικαίωμα στην ζωή είναι το πιο σημαντικό. Δεν υπάρχει πιο ουσιαστικό θεμελιώδες δικαίωμα. Και δεν θα πρέπει να κάνουμε στους άλλους αυτό που δεν θέλουμε δεν θέλουμε να συμβεί σε εμά. Και να σημειώσω ότι ο κόσμο δεν θα είχε γνωρίσει τον Πετόβεν αν η μητέρα του είχε ακολουθήσει τι συμβουλέ που τη έδιναν και είχε αποφασίσει υπέρ τη άμπλωση. Θα ήθελα λοιπόν στις αποφάσεις μας, στις δηλώσει μας να λαμβάνουμε υπόψη και αυτή την αρχή της προσοχή. Και αυτό ισχύει για όλα τα μέλη της κοινωνίας μας, ότι όλοι μπορούν να αποφασίζουν και ιδιαίτερως να αποφασίσουμε για αυτούς που δεν μπορούν να λάβουν τις δικές τους αποφασίσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να αναφερθώ στο δικαίωμα της ζωής. Όλα αυτά τα δικαίωματα τα οποία συζητάμε αφορούν και γυναίκες και α, Αλλά συχνά στις περιπτώσεις που συζητούμε δεν υπάρχει ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών. Αυτό το βλέπουμε στο επίπεδο του νοικοκυριών, σε εθνικό επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα πρέπει λοιπόν να το τοποθετηθούμε. Αλλά αυτό θα πρέπει να επηρεάσει όλους τους τομείς. Φυσικά κάτι τέτοιο θα ήταν ε, δύσκολο να το εξετάσουμε και το αποτέλεσμα του τελικό ενδεχομένω να είναι απευκταίο. Στην πρόταση του κυρίου Ταραμπέλα. Βλέπω ότι έχει ευρύ πνεύμα, ε, ακολουθεί μια σόφρυνα τακτική και υπογραμμίζει τα προβλήματα τα οποία είναι σημαντικά για τη σημερινή εποχή. Αυτό δεν σημαίνει ασφαλώς ότι δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα πέρα από αυτά. Δεν σημαίνει ότι οι γυναίκες δεν ε, αντιμετωπίζουν και άλλα προβλήματα. Εγώ λοιπόν είμαι υπέρ της διαστρωμένης ε, κατάρτισης της έκθεσης και να μείνουμε στα προβλήματα που ανέφερε εξ αρχής ο Μάρκ. Θα γνωρίζετε ότι θα αναφερθώ ασφαλώς και στο σημείο 7. Όχι από ιδεολογική άποψη, αλλά για πολιτικούς σκοπούς και μάλιστα νομοθετικού σκοπούς ιδιαίτερω. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσαν το τρέχον έτος μία δήλωση και λάβαν μία απόφαση σε ό,τι αφορά την προστασία της ζωής, σε ό,τι αφορά την υγειονομική περίθαλψη και την ανατροφή, ότι όλα αυτά ε, εμπίπτουν στον τομέα δαρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι της, ε, των κρατών μελών, και όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δικαίως είπε η συνάδελφος από την Ισπανία ότι χαίρεται που η Ισπανική κυβέρνηση απέσυρε το σχετικό νομοσχέδιο για την άμβλωση. Αλλά αυτό το αποφάσισε η Ισπανία, η Ισπανική κυβέρνηση, ο Ισπανικός λαός, όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ, Μάρκ, για το εξή. Αν δεν επιθεμεί να διχαστεί εκ νέου το Κοινοβούλιο, αν δεν θέλουμε να διακυβευτεί και η έγκριση ίδια της έκθεσης αυτής και αυτό πραγματικά δεν το επιθυμώ, γιατί για τις Ευρωπαίες γυναίκες θέλουν να εγκριθεί αυτή η έκθεση. Αν λοιπόν θέλουμε να το πετύχουμε αυτό, θα ήθελα το θέμα της άμβλωσης να παραμείνει στα χέρια των κρατών μελών και να μην ε, αναφέρεται σε θέματα που αφορούν την ισότητα. Ευχαριστώ. Κάπως δυσκολεύτηκα να τα καλύψω όλα. Αλλά πρέπει να ευχαριστήσω τον συνάδελφο για τα όσα εκείνος εκάλυψε. Και συμφωνούμε στο ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι εκείνο ασχολείται με τα ζητήματα που έχουν τι γυναίκε. Να μην τα επαναλάβω πάλι, γιατί το κατά 90% όλοι εδώ πέρα ε, συμφωνούμε, δεν είναι θέμα ιδεολογίας όταν μιλούμε για τη βία των γυναικών, όταν συζητούμε ευτυχώς συμφωνούμε σε, για κάτι τέτοιο όσον αφορά για την ε, συμφιλίωση, για τη βία ακριβώς όπως τα είπε και η ε, Ιταλίδα συνάδελφος σε σχέση με το ότι αναβάλουμε στην άκρη την ιδεολογία και να προωθήσουμε ένα τέτοιο θέμα το οποίο μας καίει και να μην επικεντρωνόμαστε σε αυτά που μας χωρίζουν, αυτά που μας ενώνουν. Οπότε και εγώ δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω και με την κυρία Ζαμπόρσκα και με τους άλλους που μίλησαν και έχω να σας πω ότι πρόκειται για μια έκθεση ευρύτατη και ήδη από πέρσι συγκεντρώθηκε μια συνένεση γύρω από αυτό και οπότε θα πρέπει επομένω να δούμε ε, τι έχει γίνει στο παρελθόν. Είχαμε δύο εκθέσεις για την βία ε, της ε, Σβένσον και η κυρία Παρμάνοβα είχε μια δεύτερη εκθέση. Και οι δύο αυτές εκθέσεις συγκέντρωσαν συντριπτική πλουσία στο Κοινοβούλιο. Πέρασαν οι εκθέσεις, εγκρίθηκαν. Γιατί, γιατί υπήρχε συνένεση. Μα έτσι πρέπει να γίνεται για κάθε έκθεση. Και πρόκειται για κάτι το οποίο πρέπει να το κάνουμε, να προωθήσουμε δηλαδή αυτές τις ιδέες, αυτές τις εκθέσεις, όχι μόνο για τις γυναίκες, για όλη την κοινωνία. Και όταν έρθει η ώρα της ε, ακρόασης θα ρωτήσω την ε, υποψήφια επίτροπο τι γίνεται με τις ε, οδηγίες που έχουν σχέση με τα δικαιώματα των γυναικών, τι γίνεται με την προστασία των θυμάτων ε, εγκληματικών ενεργειών. Τι γίνεται με τις γυναίκες που υφίστανται πάνω προώθηση, που πάνε από τη μία χώρα στην άλλη, που ξαφνικά έχουν να ε, αντιμετωπίσουν διαφορετικό δίκαιο που τις διέπει κλπ. Επίσης, όπως είχε πει και η κυρία Παραπημάνοβα τότε, στην έκθεσή της να δούμε τι θα γίνει με την βία μεταξύ των φίλων και παρά θα πρέπει να υπάρξει μια σχετική οδηγία και μέχρι να περάσει μια τέτοια οδηγία κομισιών εμείς θα πρέπει να θέτουμε το ζήτημα. Επίσης, συναρμόδια με μας είναι και η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Πέρσι είχαν μια έκθεση κατεβάσει για την κυβερνοβία κατά των ανηλίκων. Πολύ σημαντικό και αυτό και θα πρέπει να συνεχίσουμε το θέμα αυτό ε, να το προωθούμε από κοινού την Επιτροπή. Θα ήθελα να διαφωνήσω με την προπροηγούμενη ομιλήτρια Είπατε ότι οι γυναίκες έχουν ένα πρόβλημα και αναφέρετε ποια είναι τα προβλήματα των γυναικών αυτών. Εγώ δεν συμφωνώ. Η κοινωνία έχει ένα πρόβλημα και οι επιπτώσεις πλήττουν τις γυναίκες. Να πιστεύουμε ότι είναι πρόβλημα των γυναικών όταν δεν υπάρχουν χρήματα, όταν γίνονται βιασμοί, ε, είναι κάτι περίεργο. Είναι πρόβλημα της κοινωνίας και είναι σημαντικό να το θέσουμε αυτό και θα ήθελα να θέσω άλλο ένα σημείο σε ό,τι αφορά τις διαφημίσεις που βασίζονται υπερβολικά στο στο σεξ. το θέμα λοιπόν αυτό ε, τέθηκε και σε ένα εργαστήριο, σε μια εκδήλωση προσφάτως, γιατί οι γυναίκες χρησιμοποιούνται ως ε, προϊόν, προς πώληση και τι χάνουν εκμετάλλευσης για να πολλούνται αυτοκίνητα, μηχανές ή άλλα προϊόντα στους άνδρες. Αυτό σημαίνει και αυτός ο τομέας αλλά και πολλοί άλλοι τομείς θα ήθελα να συμπεριληφθούν γιατί ξέρουμε ότι ο τομέας αυτός τα τελευταία χρόνια έχει πάρει πραγματικά δυσάρεστες διαστάσεις. Ευχαριστώ κύριε Σεμπάστια. Eh, Ευχαριστώ κύριε Σιγητή. Όπως το θέτετε ιδιαίτερα μου άρεσε και από εκεί θα μπορούσε να έχουμε μια καλή έκθεση και να την εγκρίνει το Κοινοβούλιο. Είμαι καινούριο εδώ, ίσως είμαι κάπως αφελής, αλλά ε, σχετικά με το πρόβλημα αυτό θα πρέπει να δούμε και ποιοι είναι οι πέτοι στην βία κατά των γυναικών. Έχουμε νομοθεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν επιβαρύνουν τη βία αυτή ή την κρύβουν, την καλύπτουν έτσι. Λένε ότι είναι έγκλημα πάθους, έτσι τον τίνουν. Αυτό την δρομερή μάστιγα, αυτή τη βία κατά των γυναικών θα μπορούσαμε να την θεραπεύσουμε, αν το κρύβουμε έτσι, στους ποινικού κώδικες. Θα πρέπει να δούμε ε, και να θίξουμε το ότι συνεργάζονται ουσιαστικά σε αυτό το έγκλημα αυτές οι κυβερνήσεις, έτσι. Νομίζω ότι είναι σημαντικό λοιπόν να μπει αυτό το πράγμα, ότι πολλοί ουσιαστικά ε, συνεργάζονται, το ευνοούν. Τελειώσαμε με αυτό το θέμα και τώρα να δούμε τη σχόλια της Επιτροπής. Κύριε Λούσιντε Βόιλ. Euh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Γρήγορα, γρήγορα, εισαγωγικά, η αιτήσια έκθεση Επιτροπής ε, είναι για μας σημαντική δημοσίευση, δημοσίευση κλειδί για τη βία των γυναικών ε, και παρουσιάζεται ότι έχει γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτική, νομοθετική πρόοδος ε, και κάνει ένα απολογισμό του τι πρόοδος έχει επιτευχθεί σχετικά με τις προτεραιότητες και βάσει των δικτών που υπάρχουν. Το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι σε περισσότερους τομείς για τη στρατηγική υπήρξε πρόοδος, δεν είναι όμως ίσες από ένα κράτος στο άλλο και είναι και αργές και διαφέρουν από το ένα τομέα στον άλλο. Α, λοιπόν, ε, πολύ αργά προχωράει το πράγμα στις ίσες αμοιβέ. Ε, θα πρέπει να περιμένουμε ακόμα 70 χρόνια να συνεχίσουμε τον ίδιο ρυθμό το σημερινό. Με την έκθεση αυτή, με την ευκαιρία, τονίζουμε τις ε, διαφορές που υπάρχουν για τις ευκαιρίες ανάμεσα άνδρες και γυναίκες. Δεν θα υπενθυμίσω όλους τους αριθμούς των στατιστικών, τα ξέρετε, τα συζητήσατε μόλις. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα σχόλια πάντως ευχαριστώ. Και ο κύριος Αραμπέλα λοιπόν έχει τώρα το λόγο. Κύριε Αντιπρόεδρε, μετά από όσα ακούσαμε μου φαίνεται πως θα τραβήξει πολύ περισσότερο η εκθέση αυτή. Σίγουρα δεν είπα τα πάντα λεπτομερώς, έτσι. Είπα απλώς την ε, βασική διάρθρωση πως έχει. Ε, επικέντρωσα το ενδιαφέρον μου σε 7 σημαντικά σημεία που θα πρέπει να θίξουμε. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε κι άλλα. Έτσι, ε, πάντως όσα άκουσα τα σημείωσα και θα μπορούσαν να περιληφθούν ε, σε ένα κεφάλαιο ή να ανοίξουμε καινούρια. Και ας πούμε το θέμα και των συντάξεων και των ανισοτήτων στις αμοιβέ. Έτσι και τη συντάξη, όπως είπαμε που επηρεάζει τα ηλικιωμένα άτομα και το δημόσιο τι μπορεί να κάνει το δημόσιο, το δημόσιο δεν αφιερώνει πια ιδιαίτερα κονδύλια λόγω αυτής της λιτότητας ε, ή της ακραίας λιτότητας όπου εφαρμόζεται στις διάφορες χώρες. Η κυρία Ζινάσκα είπε κάτι που με απασχολεί επίσης και ο κύριος Σεμπαστιάν τώρα στο τέλο. Σεμπαστιά, Σεμπαστιά, όχι Σεμπαστιάν, Σεμπαστιά, ναι. Λοιπόν, θα πρέπει να το προσέξουμε. Καταλαβαίνω ότι σας απασχολεί να υποφεληθούμε από τις βέλτιστες πρακτικές στην Ευρώπη γιατί αρκετά κράτη έχουν προχωρήσει ιδιαίτερα και μια στιγμή δόθηκε στην Ισπανία μάχη για τη βία των γυναικών και πρέπει να το αντιμετωπίσει κανείς υπό Ισπανική Προεδρία στην αρχή από το Κάντιξ μας ε, ήταν η αρμόδια υπουργό μας τα είπε αυτά, θα πρέπει να το προσέξουμε αλλά μην δείξουμε και πεντακάθαρους μενες χάρες, ε, χώρες, ξέρετε τι σημαίνει αυτό, γιατί ε, ίσως ορισμένοι συνάδελφοι ε, θα υπεραμεινθούν λέγοντας ότι εντάξει ναι μεν το κάνουμε αυτό, αλλά προσέχουμε άλλος ε, με τη Σλοβακία λοιπόν και να προσέξουμε να μην μπούμε σε θέματα εθνικής πολιτικής ενώ μια κάποια στιγμή θα πρέπει να το λέμε και μάλιστα θετικά ποια είναι τα παραδείγματα πολιτικής που έχει ασκηθεί και αυτό ώστε να αποτελέσουν παραδείγματα καλής πρακτικής Ξέρω ότι θα υπάρξουν αντιρρήσεις όσον αφορά την άβλωση και την αντισύλληψη. Η κυρία Ζαμπόρσκα, ναι, η κυρία Λούλιν ήταν ε, το 2009 από το ΕΛΚ. Το ίδιο ακριβώς είπε. Τέλο πάντων θα συντάξω την έκθεσή μου, άκουσα τις υποδείξεις σας, αλλά δεν θέλω να μειώσω, να αφαιρέσω ε, και το είχα πει και στην κυρία Λούλιν Προτιμώ να απορριφθεί η έκθεσή μου παρά να επιμείνω στα σημαντικά θέματα. Κάτι που θα είναι πολύ ε, αποψηλωμένο, δεν θα προσέξει πολλά και διάφορα. Πρέπει να συμπεριληφθούν, δεν κάνω κάτι τέτοια. Είναι ανοιχτή πάντως η συζήτηση, ανοιχτός και εγώ και σίγουρα πάρα πολλές τροπολογίες. Θα προσπαθήσω να βρω σίγουρα τέτοιος τύπος είμαι ε, μια συνένεση και θα προσπαθήσω να προχωρήσω στις συμβαστικές λύσεις, να μπορέσω να λάβω υπόψη μου διάφορες τροπολογίες, να μην λάβω υπόψη με άλλες. Θα πρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στείλουμε ένα μήνυμα που να υπογραμμίζει, να τονίζει τα δικαιώματα των γυναικών, επίσης όμως και τις ελλείψεις στα διάφορα προβλήματα που ισχύουν σήμερα και να προτείνω και λύσεις. Σας ευχαριστώ για την προσοχή που με αφιερώσετε, δεν μένει παρά να σκουμποθούμε και να ρηχτούμε στη δουλειά. Ευχαριστώ κύριε Μαγκαραμπέλα. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Όσον αφορά το άρμα πρόδια των γυναικών. Οι συνεργαστές πάνε να θα πρέπει να υπάρξει κάποιο ψηλό επίπεδο διάσκεψη ε, και να γίνει κατά την συνάντησή μας του Νοεμβρίου. Κύριε Ντάγμαρ Σουμάχερ, παρακαλώ, παρουσιάστε μας τις λεπτομέρειες για αυτήν την ε, διάσκεψη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ντάγμαρ Σουμάχερ, με μεγάλη μου χαρά είμαι εδώ και είμαι διευθύντρια του γραφείου του ΟΗΕ εδώ στις Βρυξέλλες. Είναι πρώτη φορά που έρχομαι στην ε, ε, Επιτροπή της Νέας Θητείας, οπότε σας εύχομαι ότι καλύτερο και ευχαριστούμε να συνεργαστούμε μαζί σας στους αμέσως επόμενους μήνες. Όσον αφορά τώρα αυτό το άλλο πρόοδο, είναι πάρα πολύ σημαντικό και μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προχωρήσουμε. Τον Οκτώβριο του 2012 υπεγράφει ε, ε, η σχετική πρόταση και Είχαμε ήδη συνεχθεί από αυτού με την Επιτροπή Γενικών της τελευταίας κοινοβουλευτικής θητείας. Τώρα, αυτό το οποίο θέλουμε είναι να γίνει μια διάσκεψη υψηλού επίπεδου, 5 και 6 Νοεμβρίου. Τι σημαίνει άλμα πρόοδου. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο εξετάζει την οικονομική και πολιτική συμμετοχή των γυναικών στην Αραβία. Έτσι έχουμε αυτή τη διάσκεψη ε, υπό την ηγίδα της Επιτροπής ε, Γυναικών. Έχουμε τώρα τις ημερομηνίες, έχουμε τα σχετικά μηνύματα, ε, μας βοήθησε στη, στις σχετικές ειδοποίησεις και προσκλήσεις η γραμματεία σας και ευχαριστούμε και θέλουμε τελικά να καταλήξουμε σε κάποιο είδους δίκτυο για ανταλλαγή εμπειρίας, και έτσι να υπάρξει τελικά μια συνένεση για τα θέματα της ισότητας των φύλων και αποτελεσματικής ηγεσία ε, και αυτό να διαμορφωθεί μεταξύ των ευρωβουλευτών και των ε, βουλευτών των χώρων που αναφέραμε. Έχουμε περίπου 30 με 35 γυναίκες που νομοθετούν και θα έρθουν σε αντιπροσωπεία και έρχονται από Αραβία, Μαγρέμπ, Μασρέκ, Ιράκ και Παλαιστίνη. Έχουμε δύο με τέσσερις εκπροσώπους αναχώρα. Βεβαίως, η στενή συνεργασία με ε, αυτούς που θα έρθουν είναι πάρα πολύ θετικό. Σε σχέση με αυτή την εκδήλωση ελπίζουμε να έρθει και ο Μαρτίν Σούλτς, ο πρόεδρος, να έρθει ο εκτελεστικός διευθυντής ε, του ΟΗΕ για τις γυναίκες, ίσως ε, ο ή επίτροπος τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίσης ε, κάποιος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής ε, Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Θα προεδρεύσει η Πρόεδρος Επιτροπής Γυναικών. Την πρώτη μέρα, στις 5 ε, Νοεμβρίου του 2014, θα εξετάσουμε ζητήματα, προκλήσεις και ευκαιρίες όσον αφορά τη συμμετοχή των γυναικών. Όσον αφορά το mainstreaming, τη ισότητα για τις εθνικές νομοθεσίες, για το πώς θα συμμαχήσουν οι γυναίκες προς την νομοθεσία σε σχέση με τα μίντια και τις ε, οργανώσεις διάφορους φορεί Οπότε γι' αυτό και θέλουμε τα μέλη της αντιπροσωπείας κάθε πρόσφυγη που θα έρθουν ποια πιο σημαντικά ε, θέματα ούτως ώστε να μπορέσουμε και εμείς να προσαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Επίσης και το Ευρωκοινοβούλιο ε, αν θέλει μπορεί να υποδείξει το ποια θέματα επιθυμεί να συζητηθούν. Τη δεύτερη μέρα τώρα τις διάσκεψης τα μέλη της αντιπροσωπείας τραβούν μέρος σε συναντήσεις με το Κοινοβούλιο ε, κάπως πιο άτυπα από την πρώτη μέρα. Επίσης, στο ξενοδοχείο θα έχουμε ένα ε, δείπνο, γεύμα και όλοι μπορείτε να προσέλθετε. Είστε καλεσμένοι. Αυτά είναι μια πολύ μικρή σύνοψη και βεβαίω ό,τι ερώτηση έχετε μπορείτε να την ε, υποβάλλετε. Και φυσικά χαιρετίζω το πόσο ζεστά πήρατε αυτή την εκδήλωση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, Ντάκμαρ Σούμαχερ. Συνάδελφοι, αν έχετε ερωτήσεις, παρατηρήσεις για το συνέδριο αυτό, παρακαλώ να τις θέσετε. Όχι, δεν υπάρχουν ερωτήσει. Μάλιστα, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε την κυρία Σούμαχαρ. Σας ε... να συμμετάχετε σε αυτή τη διαδικασία, σε, αυτή την, ε, σε αυτό το συνέδριο. Θα ήθελα να πω ότι έτσι ολοκληρώσαμε την εξετασία όλων των σημείων στην ημερήσια διάταξη στις 6 Οκτωβρίου δεν θα γίνει η συνεδρίαση και άρα η επόμενη συνεδρίαση θα λάβει χώρα στι 13 Οκτωβρίου πέρα της συνεδρίασης.